καθημερινά να ακολουθούν οι αλλοίς όταν ψαρεύουν. Γιατί θέλω να επιβάλλω αυτά τα μέτρα στους ε, αλλοίς για να διασφαλίσουμε ότι η αλληλεία γίνεται με βιώσιμο τρόπο. Αυτή είναι η κόκκινη γραμμή της έκθεσής μου. Βιωσιμότητα. Καταλαβαίνω την αναγκαιότητα των μέτρων αυτών, ούτως ώστε τα αποθέματα να αλλιεύονται με βιώσιμο τρόπο και τα οικοσυστήματα στα οποία ζουν τα ψάρια να διατηρούνται. Για να είναι αποτελεσματικά αυτά τα μέτρα και να επιτύχουμε τους στόχους μας, τα μέτρα αυτά πρέπει να διατυπωθούν λαμβάνοντας υπόψη την εξελικτική φάση, ε, φύση της αλίας και με επιστημονικές συμβουλές. Εάν δεν είναι τα σωστά τεχνικά μέτρα, εάν δεν τα ε, εκπονήσουμε σωστά, μπορεί να έχουμε μη βιώσιμες ε, πρακτικές αλίας που να θέσουν εγκυνδύνο κινδύνο τη βιωσιμότητα των αποθεμάτων και να θέσουν εγκυνδύνο τη ζωή και ασφάλεια και των αλλοίων μας. Κάτι που θα ήταν απόλυτα απαράδεκτο. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα. Είχαμε μια έκθεση σήμερα το πρωί που εγκρίναμε για την μικρή κλίμακα και παράκτη αλλοία ή αλληλείς. Ε, εργάζονται σε πολύ σκληρές συνθήκες. Πρέπει λοιπόν να τους προστατεύσουμε. Υπάρχουν κάποια ε, μέτρα για τον περιορισμό της αλίας, του γάδου και του φαγκριού έχουν να κάνουν με το η περιοχή όπου γίνεται αυτή η αλία δεν είναι η, η πρέπουσα. Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν τεχνικά μέτρα τα οποία τα χρειαζόμασταν και όταν εγκρίναμε τον βασικό κανονισμό της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Είναι επίσημα σημαντικό να σημειώσουμε ότι τα μεταβατικά τεχνικά μέτρα τα έχουμε εδώ από την 1η πρώτου 10. Ισχύουν δηλαδή από τότε, όπως όλοι ξέρουμε, λίγουν τέλος του χρόνου. Είναι λοιπόν ουσιώδες να πάρουμε απόφαση εάν θα προσπαθήσουμε να καταλήξει αυτή η έκθεση πριν τέλος του χρόνου, ουσιώδε να παρουμε αλλιώς θα πάψουν να ισχύουν τα προσωρινά μέτρα. Η Κομισιόν θα μπορούσαν για άλλο 1,5 χρόνο να παρατείνουν την ισχύ τους. Δύο φορές έχει υπάρξει αυτή η παράταση των προσωρινών μέτρων. Προτείνουν να τροποποιήσουν λοιπόν τον αρχικό κανονισμό 88-50 του 88. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν θα έχουμε όλα τα βασικά στοιχεία της μεταρρύθμισης της κοινής ελευθερικής πολιτικής πριν το 2015. Είναι πολλά, λοιπόν επιτακτικό τα προσωρινά μέτρα που αντιβαίνουν τη βιωσιμότητα των αλλιευμάτων να τροποποιηθούν. Αυτό δεν είναι μόνο κοινή λογική, είναι υποχρέωσή μας έναντι των εκλογέων. Τα μέτρα βασίζονται σε συγκεκριμένα άρθρα και επιχειρούν να τα απαλείψουν. Γιατί ορισμένα από αυτά είναι πλέον πεπαλαιωμένα. Και υποστηρίζονται οι προτάσεις μου, τονίζω, πλήρως από τους επιστήμονες. Πολλά από τα προβλήματα που έχουν αυτή τη στιγμή οι μας, για παράδειγμα ο τομέας IC6A, έξω από την ε, δυτική ακτή της και τη βορειοδυτική ακτή της Ιρλανδίας, έχουν να κάνουν με τον αρχικό κανονισμό. Όλοι λοιπόν πρέπει να συμμετάσχουν. Θα το συζητήσουμε και αλλού. Είναι λοιπόν χαρακτηριστικό παράδειγμα επειδή είναι πήγο το θέμα έχω συμπεριλάβει και τροπολογίες που θα σας εξηγήσω σύντομα. Αν αναγκαίο μπορώ να τις κάνω τροπολογίες. Τροπολογίες 1 και 3 είναι τεχνικές. Έχουν να κάνουν μόνο με το που πρέπει να πάνε οι αιτιολογικές σκέψεις 9 και 11. Και οι δύο ανταποκρίνεται στην ανάγκη να διορθώσουμε ένα λάθος. Οι 4, 5 και 6 έχουν να κάνουν με τις απορρίψεις και την υποχρέωση να ε, φτάνουν στην ακτή όλα τα λιεύματα. Και τώρα θέλω να βάλω στον κανονισμό ένα νέο άρθρο και είναι μόνο προσωρινό. Θα πρέπει λοιπόν να περιμένουμε την έγκριση του βασικού κανονισμού. Πιστεύω ότι η Επιτροπή, καλή την πίστη πιστεύω, προσπαθούν να προλάβουν, να προκαταλάβουν τις ε, διαπραγματεύσεις μεταξύ μόνο και του Συμβουλίου. Η Κομισιόν λοιπόν θα φέρει ένα νέο κανονισμό, θα υποβάλει ένα νέο κανονισμό μετά τον βασικό κανονισμό της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Ο νέος κανονισμός και όχι αυτός ο προσωρινός κανονισμός είναι ο καλύτερος για να αναφερθούμε στην ανάγκη να φτάνουν στην ακτή όλα τα λεύματα. Έχουμε και άλλες σημαντικές τροπολογίες γιατί πρέπει, όπως λένε οι επιστήμονες, να αλλάξουμε τους ε, καθορισμένους χώρους αλίας. Λαμβάνω υπόψη λοιπόν τις ε, οδηγίες του Οι 7 αλλάζει την κατάσταση της γραμμής και η 15 λέει ότι μπορεί να πάει να ε, κινηθεί περαιτέρω ή και να παλευθεί χωρίς να χρειαστεί να επανέλθει το κοινοβούλιο. Άλλη τροπολογία έχει να κάνει με τους αλληλείς μικρής κλίμακας που εργάζονται με πολύ σκληρή συνθήκη στον Ατλαντικό. Δεν χρειάζεται να εξαιρούμε κάποιο είδος εξοπλισμού που χρησιμοποιούν Σήμερα εγκρίναμε την έκθεση για τη μικρή κλίμακα αλληλεία. Δεν θα ε, μπω σε αυτό το θέμα. Απλώς πρέπει να τονίσω ότι έχει πολύ θετικές συστήσεις. Οι 10, 11 και 13 αναγνωρίζουν ότι έχει υπάρχει έκρηξη του, του γάδου και γι' αυτό έχει ε, βγει από τον κανονισμό για τα παράπλευρα αλλιεύματα εκπλήσουμε που η Κομισιόν δεν έδρασε με το θέμα αυτό. Η 12, μάλλον η 14 έχει να κάνει με τις απορρίψεις και την προστασία του γόνου και θα προτείνω μερικές περιοχές όπου θα απαγορεύεται η αλίευση. Αυτό είναι ίσως περίεργο που το κάνει ένας Ευρωβουλευτής, αλλά στη χώρα μου υπάρχουν ήδη. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσουμε να συνεργαστούμε Σύντομο θα είναι το διάστημα για υποβολή τροπολογιών, αλλά ίσως ε, χωρίς να θέλω να προκαταλάβω την εργασία σας, να μην χρειάζονται και τόσο πολλές τροπολογίες στην εκθεσή μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ταχύτητα. Έχουμε μόνο πέντε λεπτά. Ίσως και λίγο χρόνο παραπάνω που θα μας δώσουν ε, οι διερμηνείς, ίσως 10 το πολύ. Τέσσερις έχουν στήσει το λόγο. Ένα λεπτό παρακαλώ, ούτως ώστε μετά να κλείσουμε το θέμα η κυρία Ντότς πρώτη παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να τηρήσω το χρονικό όριο. Όπως συνήθω με τις ε, παρεμβάσεις του ΠΑΤΑΚΟΠ είμαι υπέρ αυτής της έκθεσης, ωστόσο υπάρχει μια τροπολογία που με απασχολεί και με ανησυχεί, η 14, που προβλέπει την εισαγωγή ενό ε, κλεισίματο περιοχής για έξι μήνες για οποιασδήποτε αλληλευτικές δραστηριότητες με εξοπλισμό που αν φέρονται στο παράρτημα 1 του κανονισμού 1342 του Συμβουλίου διάφοροι εξοπλισμοί που στοχεύουν σε είδη βυθοβία τα οποία εξετάζονται για εξαίρεση από το μακροχρόνιο σχέδιο είτε λόγω της τροποποίησης των εξοπλισμών ή στην περίπτωση των εξοπλισμένων άλλων διότι έχουν παρεπίπτοντα λιεύματα. Αυτή τη στιγμή προτείνουμε λοιπόν ε, ε, προσωρινό κλείσιμο για αυτά τα ήδη. Θα θέλαμε λοιπόν να το συζητήσουμε. Ευχαριστώ. μας παρακαλώ. Oui, merci, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι και εγώ σύντομη. Συμμερίζομαι τις απόψεις του εισηγητή. Μου αρέσει που μένει πιστό στην επιστημονική διαδικασία, ειδικά όταν μιλάει για τα αλλιευτικά εργαλεία, αλλά και για την επιτήρηση για, και τη μέρημνα για βιώσιμη αλληλεία. Συμφωνώ επίση μαζί του στο γεγονό ότι ακόμη και αν είναι καλόπιστη η Επιτροπή, δεν χρειάζεται να προβλέψουμε τι θα αποφασιστεί για τι εκφορτώσει αλλιευμάτων και να απομακρυνθεί όλο αυτό από τον κανονισμό. Επίσης, συμφωνώ μαζί του, πρέπει επίγοντα τα επίγοντα μέτρα να γίνουν μεταβατικά, διότι δεν μπορούν να αναμένουν την ψήφιση του βασικού κανονισμού, κυρίως γιατί δεν ξέρουμε πότε θα λάβει η χώρα. Θα ήθελα να τονίσω ότι ακόμα μελετώ και άλλες επίγουσε καταστάσεις, πιθανές. Νομίζω ότι έχουμε μέχρι την Παρασκευή για τις τελευταίες τροπολογίες. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να τροφοδοτήσουμε ακόμη περισσότερο την έκθεση του κ. Γκάλαχερ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Χάρτον και εσείς ένα λεπτό. Thank you. Um, difficult in one minute, cause it's... Είναι δύσκολο σε ένα λεπτό γιατί είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα και μιλήσαμε ελάχιστα γι' αυτό. Η κατάσταση εδώ έχει ως εξής η Κομισιόν για κάποιο λόγο δεν χρησιμοποιεί πρακτικά μέτρα σε μια κατάσταση όπου έχουμε δύο πράγματα που και όλοι βλέπουμε ότι δεν θέλουμε να κάνουμε. Ε, το να απορρίπτουμε τα καλά ψάρια και το να μην συμμορφωνόμαστε με τους κανονισμούς. Για να μειώσουμε τις απορρίψεις του γάδου στη Δυτική Σκοτία όπως αναφέρεται από τον ε, εισηγητή παρότι έχει αναγνωριστεί το γεγονός και έχουν γίνει δεκτά τα επίγοντα μέτρα και έχουν ελοπεωθεί για να αντιμετωπιστεί αυτό το γεγονός, παραμένουν οι αιτίε των απορρίψεων και αυτή τη απαράδεκτη κατάσταση, όχι μόνο για του αλλοί αλλά και μια παράλογη κατάσταση. Δεδομένων των όσων λέμε εδώ πέρα για τι απορρίψει ε, και για τη μείωσή του. Εδώ έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να δείξουμε ότι το εννοούμε όταν λέμε ότι θέλουμε το νέο καθεστώς διαχείριση τη αλληλείας να είναι πιο λογικό, πιο πρακτικό και να λειτουργεί πραγματικά και όχι απλά να είναι θεωρητικέ ιδέε. Ελπίζουμε λοιπόν ότι μαζί με τον κύριο Γκάλεχερ θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κυρία Λοβίν, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Απλά ήθελα να πω ότι θεωρούμε ότι αυτή η εκθέση είναι θεμελιώδη σημασία. Τα τεχνικά μέτρα που έλειπαν εδώ και πολύ καιρό είναι υπερβολικά σημαντική για να τη συζητήσουμε σε 14 λεπτά εντός της Επιτροπής και μετά να έχουμε προθεσμία υποβολής τροπολογιών την Παρασκευή. Προτείνω λοιπόν να παρατείνουμε την ε, προθεσμία υποβολής τροπολογιών για να έχουμε χρόνο να συζητήσουμε με τον εισηγητή και να μπορέσουμε να μελετήσουμε σε βάθος αυτή την ε, θεμελιώδη σημασία έκθεση, όπως είπε ο εισηγητής, ε, αναφέρει πολλά ζητήματα πολύ σημαντικά Θεωρούμε λοιπόν ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε να περάσουμε τόσο βιαστικά μια τέτοια έκθεση. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και τη... να παρατείνουμε και την ίδια την έκθεση και θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα την παράτηση τη προθεσμίας υποβολή Τροπολογία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα πρέπει να έχουμε και ένα λεπτό και για την Επιτροπή. Παρακαλώ να μας δώσουν πέντε λεπτά ακόμα οι διερμηνείς και υπόσχομαι ότι θα ολοκληρώσουμε μετά από αυτά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, στην Επιτροπή, ποιε είναι οι δυνατότητε ε, για την προθεσμία για τι τροπολογίε. Το περισσότερο, το μέγιστο θα ήταν την Δευτέρα στι 10 το πρωί εκνοή τη προθεσμία. Θα είχαμε και την Παρασκευή και το λίγο το, του πρωινού τη Δευτέρα. Αν συμφωνείτε σε αυτή την περίπτωση, δεν ε, κερδίζουμε και πάρα πολύ. Δεν έχουμε άλλο περιθώριο, ούτω ή άλλω μα λένε. αυτό είναι αυτό που ξέρουμε. Κύριε Γκάλαγκερ, uh, uh, Αν το δέχεται η γραμματεία, θα ήθελα και εγώ περισσότερο χρόνο. Αλλά οι προθεσμίες είναι τέτοιες που ε, εάν επιμικρύνουμε την προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών δεν θα προλάβουμε να εγκριθεί μέχρι τέλος του χρόνου. Οπότε όλη η δουλειά που θα κάνουμε θα πάει στράφη. Θα επανέλθουμε στην κατάσταση πριν από 3,5 χρόνια. Γιατί υπάρχει πίεση να επεκταθεί η χρήση των ε, προσωρινών μέτρων, η ισχύ των προσωρινών μέτρων. Δευτέρα λοιπόν ε, στις 10 το πρωί, ούτως ώστε να έχετε σαν το Κυριακό. Να ακούσουμε και την Κομισιόν ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Σε ένα λεπτό τώρα τι σχόλια να κάνω. Θα επιχειρήσω όσο πιο σύντομο γίνεται. Ευχαριστούμε και τον εισηγητή για την ταχύτητα με την οποία ε, Παρουσία στην έκθεση που σχετίζεται με το πολύ αυστηρό χρονοδιάγραμμα που έχουμε ούτως ώστε να παραμείνουν αυτά τα τεχνικά προσωρινά μέτρα. Μέχρι το τέλος του χρόνου λοιπόν πρέπει να εξετάσουμε το θέμα αυτό. Άκουσα ότι ίσως να υπάρχουν αμφιβολίες και κάποιες έννοιες που μπορούν να βοηθήσουμε να διευκρινιστούν. Ε, η τροπολογία 4 για παράδειγμα. Δεν προσπαθούμε να προκαταλάβουμε τις συζητήσεις στα πλαίσια της μεταρρύθμισης. Ε, διατηρούμε την απαγόρευση που υπάρχει από το 2009. Δεν είναι λοιπόν ε, καμία προσπάθεια προκατάληψης για την απαγόρευση των απορρίψεων. Αλλά μπορούμε και γραπτά να σας δώσουμε εξηγήσεις για την τεχνική φύση αυτού του θέματος για να βρούμε τον καλύτερο τρόπο για την επιστημονική, ε, επιστημονικές συμβουλές, συμβουλές που λαμβάνουμε. Είπαμε ότι θέλουμε να βασιζόμαστε πάντα στις επιστημονικές συμβουλές. Άρα για την τροπολογία 7, ίσως θα έπρεπε να συζητήσουμε με τον κύριο Γκάλεχερ την επιστημονική βάση της τροπολογίας που προτείνει, γιατί εμείς ε, Φαίνεται ότι έχουμε διαφορετικής, διαφορετικής φύσης ε, συμβουλές από τους επιστήμονες. Και τέλος, για την ε, εξαίρεση του, του μπακαλιάρου, του μελανόγραμμου γάδου από τα μέτρα αυτά. Για τεχνικούς λόγους το προτείνουμε. Τα ε, πήγοντα μέτρα ήταν για να αντιμετωπίσουν επίγουσες καταστάσεις που είχαν συγκεκριμένη χρονική ισχύ. Αν ε, τα προσωρινά ε, αυτά μέτρα θέλουμε να τα κάνουμε μόνιμα, θα είχαμε πρόβλημα νομικής αντίφασης. Προσπαθούμε φυσικά να μείνουμε στην ίδια λογική και το συζητήσαμε στο Συμβούλιο με τα κράτη-μέλη, αλλά θέλουμε να καταλάβετε ότι νομικά δεν έχουμε άλλη επιλογή, ε, όσο και αφαίνεται παράλογο. αλλά ε, με καλή διάθεση να εξετάσουμε τι δυνατότητες θα είχαμε. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά φυσικά είμαστε στη διάθεσή σας για να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Οπωσδήποτε θα υπάρχουν περιπτώσεις όπου θα το συζητήσει το θέμα αυτό με τον κύριο Γκάλαχαρ. Θα διατηρήσουμε λοιπόν την προθεσμία για τις τροπολογίες 21 12 το μεσημέρι, 21 Σεπτεμβρίου 12 το μεσημέρι, δεν αλλάζει τίποτα. Θα μείνει όπως είναι η προθεσμία. Στις 21 λοιπόν, 12 το μεσημέρι, Παρασκευή 21 Ενάτου. Εντάξει, ωραία. Κυρία Λόβιν. Μα είπαμε μέχρι τη Δευτέρα έτσι, δεν είπατε. 10 η ώρα. Ναι, αλλά μόλις ε, έλαβα το μήνυμα ότι δεν είχατε πρόβλημα εσείς. Έτσι άκουσα. Μου ανάφερα το όνομά σας. Όχι. Εντάξει, ωραία. Δευτέρα, Δευτέρα, Δευτέρα. Ε, έτσι κατάλαβα, έτσι κατάλαβα, δεν το επινόησα. Δευτέρα 10 το πρωί. Λίγη η προθεσμία υποβολής τροπολογιών. Εντάξει. Οπότε διακόπτουμε παρακαλώ. Δευτέρα λοιπόν στις 10 εκπνέουν οι προθεσμίες για τις τροπολογίες. Θα ξεκινήσουμε ακριβώς λοιπόν στις 3 ε, και κλεισμένο το θυρών. Να είσαστε στην ώρα σας εδώ. Γεια.